at this moment. Uh, I'm sure that will evolve as, uh, as we progress. But... Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ε, καλωσορίσω στην συνεδρία συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα. Μίχαελ, καλώς ήρθες. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων λοιπόν με τον Βιτσέντζο Κοπόλη, ο οποίος είναι διοικητής μη στρατιωτικών επιχειρήσεων και διευθυντής του CPCC από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και εξ ονόματος της υποεπιτροπής μας θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Είστε ο νέος διοικητής λοιπόν των μη στρατιωτικών επιχειρήσεων και διευθυντής του CPCC. Ο διορισμός σας έλαβε χώρα σε μία αρκετά δύσκολη και, αλλά και ενδιαφέρουσα εποχή. Τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να δώσουν όθηση και να ενισχύσουν τις νέες αποστολές. Και το Νοέμβριο του 2018, στην προηγούμενη συζήτησή μας, ε, μιλήσαμε για τη νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση και το εσωτερικό και εξωτερικό πλέγμα και συνεργασία ανάμεσα σε μη στρατιωτικέ και στρατιωτικέ επιχειρήσεις. Η κατάρτιση και η πρόσληψη εμπειρογνωμόνων είναι αναγκαίες έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ε, έγκαιρη ανάπτυξη ε, των ε, διαφορών δυνάμεων και επιχειρήσεων. Και επιπλέον οι αστυνομικές αρχές σε συνεργασία με τις με την ε, δημοσιοδίκηση θα αναλάβουν νέα καθήκοντα που έχουν σχέση με την ε, παράτυπη μετανάστευση που όπως γνωρίζετε είναι ένας ε, τομέας που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις κυβερνοαπειλές, την τρομοκρατία και τη ριζοσπαστικοποίηση, το οργανωμένο έγκλημα, την ασφάλεια σε ξηρά και θάλασσα αλλά και την αντιμετώπιση του βίου εξτρεμισμού και την προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς. Όλα αυτά λοιπόν είναι καθήκοντά σας, είναι πάρα πολύ σημαντικά και για εσά αλλά και για την Επιτροπή μας. Γι' αυτό λοιπόν πριν την έγκριση της συμφωνίας, τα κράτη-μέλη έχουν ζητήσει την έγκριση ενός σχεδίου στρατηγικής, το οποίο θα ε, συντονίζει δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι έχουν εκφράσει την βούληση τους να συμμετέχουν συμμετάσχουν σε αυτή, αυτό το εγχείρημα. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε από εσά να μας παρουσιάσετε το μέλλον της συνεργασίας με το Κοινοβούλιο και πώς ε, εμείς μπορούμε να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη του, ε, της κοινή ε, πολιτικής ε, ασφάλειας και άμυνας και την διεύρυνση των μη στρατιωτικών επιχειρήσεων για παράδειγμα πρόσφα... και καθώς και την επέκταση του σε βάθο χρόνου. Πρόσφατα αρκετέ αποστολέ πήραν παράταση της εντολής του και χρειάστηκαν τροποποίηση έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν διάφορε άλλε προκλήσει όπω η παράτυπη μετανάστευση, λαθρεμπόριο και τα λοιπά. Θα ήθελα λοιπόν μετά από αυτήν την ε, σύντομη εισαγωγή να δώσω το λόγο στον ε, κύριο Βιτσέντσο Ευχαριστώ. Πήρατε τα λόγια το στόμα μου. Διάφορα πράγματα από αυτά που είπατε σκόπευα να τα πω στην παρουσίασή μου. Ή τουλάχιστον θα τα θέσω επιτάπητος ε, για να τα έχουμε υπόψη όλοι. Yes. Um, yes, as you said, I started my... Ξεκίνησα το Σεπτέμβριο του 2018, ανέλαβα το πόστο μου. Η προηγούμενη θέση μου ήταν ε, ε, αναπληρωτής επικεφαλής των Καραμπινιέρη στην ε, Ιταλία. Ε, όμως όταν ξεκίνησε η ΚΕΠΑ, το μη στρατιωτικό σκέλο, ε, το 2001 με 2004 επίση υπηρέτησα και ήμουν επικεφαλής αποστολή στην Βοσνία για τρία χρόνια. Επομένω, χρησιμοποιώ αυτές τις παλιές εμπειρίες μου για τη σημερινή μου θέση, παρότι έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα από τότε που έφυγα το 2008. Θα ήθελα να πω δύο λόγια ε, γενικά για την ε, μη στρατιωτική ΚΕΠΑ και τις ε, αποστολές που έχουμε, τις επιχειρήσεις που έχουμε, χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα όμως να σας πω ποια είναι η άποψή μου. Ε, η σημερινή μη στρατιωτική ΚΕΠΑ είναι πολύ σημαντική και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται πολύ αποστολέ που έχει επιτόπου γιατί είναι ορατές, αποτελεσματικές, επιχειρησιακές, παρούσες με μια εντολή, με πόρους επαρκής για να μπορέσουν να επιδράσουν ε, σε τοπικό επίπεδο με τις τοπικές αρχές στις χώρες όπου τις έχουμε αναπτύξει και μπορούν να επιτύχουν ε, πραγματικά αποτελέσματα. Φυσικά υπάρχουν διαφορέ, υπάρχουν στο είδος αποστολής, στο μέγεθος της ε, αποστολής, ε, στην εντολή, στην διάρκεια της ε, αποστολής και της επιχείρησης. Όλα αυτά επηρεάζουν το επιχειρησιακό δυναμικό της αποστολής. Αλλά με βάση τα σημερινά δεδομένα και με την προβλεπόμενη αύξηση, αύξηση των πόρων και του προσωπικού κάποιων αποστολών, το επιχειρησιακό μας δυναμικό συνολικά θα αυξηθεί. Όλα αυτά ήθελα να τα επενθυμίσω. Να υπενθυμίσω μία έννοια που δεν πρέπει να ξεχνάμε, που είναι ε, η μελλοντική ασφάλεια ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπήρχαν και στα έγγραφα του Σολάνα για μια καλύτερη Ευρώπη και μια ασφαλή Ευρώπη σε ένα καλύτερο κόσμο, θα θυμάστε λέγαμε τότε. Στην στρατηγική ασφαλείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μιλάμε για αποστολές ε, σε σημεία κρίση και αυτό είναι τρόπος για την Ευρώπη για να εξασφαλίσει, να έχει κάποια εργαλεία ασφάλειας. Ε, η μη στρατιωτική ΚΕΠΑ και το σύμφωνο της, για την ΚΕΠΑ, της, το, του μη στρατιωτικού σκέλου. Υπάρχει ένα στρατηγικό έγγραφο που μιλάει για τη δέσμευση των κρατών μελών να αυξήσουν την παρουσία τους ε, μέσω της αποστολής να δώσουν ε, περισσότερους πόρους, ανθρώπινους πόρους κυρίως, μαζί με το πολιτικό πλαίσιο και την υποστήριξη που θα δώσουν, αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τα κράτη-μέλη, παρότι είναι το μεγάλο κομμάτι, αφορά και τα, το θεσμικό επίπεδο, γιατί η δέσμευση των κρατών μελών συνοδεύεται από διάφορα μέτρα από πλευράς μας, από την μη στρατιωτική ΚΕΠΑ, την CPCC, δηλαδή τη μη στρατιωτική δυνατότητα σχεδιασμού και διεξαγωγή επιχειρήσεων, για να διαχειριζόμαστε αυτού του πόρου ε, που θα αναπτυχθούν στο εγγύ μέλλον. Υπάρχει δέσμευση να φτάσουμε στο 100% του δυναμικού μας το 2023. Θα είμαστε έτοιμοι δηλαδή να συνοδεύσουμε τότε αυτά τα μέτρα με τα δικά μας μέτρα. Τα μέτρα των κρατών μελών δηλαδή. Το θέμα δεν είναι μόνο θέμα διαχείρισης των πόρων, αλλά είναι και θέμα καλύτερης διάθρωσης των δυνατοτήτων μας, ούτω ώστε να είμαστε καλύτεροι, σε καλύτερη θέση για να διαχειριστούμε τις αποστολές. Οι αποστολές είναι διαφορετικές. Πρέπει να έχουμε τις δυνατότητες κάθε αποστολή να διαχειριζόμαστε με βάση τις ιδιαιτερότητές της. Ε, και αυτά κάνουμε από πλευρά μα για να το πετύχουμε. Κάνουμε κάποιες, κάποια τεχνικά πράγματα. Υπάρχει το CPCC και ελπίζω το CPCC να ενισχυθεί συν χρόνο ε, με περισσότερους πόρους, όχι μόνο ανθρώπινους, αλλά και τεχνικούς. Αλλά αυτό θα το λύσουμε στο δικό μας επίπεδο με βάση τις δικές μας αρμοδιότητες. Για τις αποστολές τώρα που έχουμε... Είναι 10 συνολικά, τελείως διαφορετικές ημένα από τις ΔΕ. Πολλές, πάρα πολλές οι διαφορές. Το... Θα ξεκινήσω από την ε, πιο προβληματική περιοχή σήμερα, στη Σαχέλ. Έχουμε δύο ε, αποστολές εκεί. UCAP, Σαχίλ, Μαλή μία για το Μαλί και μία για το Νίγηρα ε, με ένα περιφερειακό πυρήνα συντονισμού για την σταθεροποίηση της Ταχέλ που θα ενισχυθεί αυτός ο πυρήνας ας πούμε και θα είμαστε θα αλλάξει τοποθεσία, θα είμαστε πολύ κοντά στη γραμματεία του DG5 για να συντονιστούμε ε, με το πολιτικό επίπεδο του G5. Οι δύο αποστολές ε, δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες, ειδικά στο Μαλή, γιατί η κατάσταση ασφαλείας στο Μαλί είναι πολύ δύσκολη. Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε ή να είμαστε μάρτυρες ε, τρομοκρατικών επιθέσεων το περισσότερο κομμάτι της χώρας ε, είναι κλειστό σε εμά. Θα πρέπει να περιορίσουμε την παρουσία μας, δηλαδή, κοντά στον Μπα, Μπαμάκο. Μπορούμε να κινηθούμε λιγάκι στο Σεγκού. Θα δούμε όμως τι θα συμβεί σύν το χρόνο. Αλλά και οι δύο αποστολές πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι που, είναι ευπρόσδεκτες από τις τοπικές αρχές Τις επισκέφθηκα και τις δύο, το αποτέλεσμα ήταν πολύ θετικό, ήμουν ικανοποιημένος και το πολιτικό και το επιχειρησιακό επίπεδο των δύο χωρών ε, επιθυμεί την παρουσία μας. Συνεργαζόμαστε πολύ με το G5, G5 και μέσα στην, ε, στην κοινή δύναμη του G5 θέλω να τονίσω την παρουσία του Συμβούλου ε, για την Αστυνομία. Ένα άτομο είναι σύμβουλος προς την τοπική αστυνομία. Θα θέλαμε όμως να πλουτίσουμε, να εμπλουτίσουμε αυτή την, αυτό το team, τέλος πάντων, το άτομο αυτό να μην είναι μόνο του. Θα το δούμε σύντομα. Στην Αφρική πάλι, μια άλλη ευαίσθητη αποστολή είναι η UCAP στη Σομαλία. Ξεκίνησαν με εστίαση στην θαλάσσια ασφάλεια. Σήμερα επεκτείνουν το δυναμικό τους ε, και τις δυνατότητές τους στο να παρακολουθούν τις αστυνομικές δυνάμεις, προσπαθούν να, ε, ε, να συντονίσουν την διμερή και την πολυμερή δύναμη που είναι παρούσα στη Σομαλία, όπου έχουμε πολύ δύσκολη κατάσταση ό,τι αφορά την ασφάλεια. Είχαμε ήδη κάποιες ε, τρομοκρατικές επιθέσεις, καμιά, καμιά δυο δηλαδή, ή τουλάχιστον κατά των διεθνών δυνάμεων και εναντίον της EUTM, μια άλλη σημαντική ευρωπαϊκή παρουσία Κάναμε κάποιες διευθυντικές αποστολές στο βορρά της Σομαλίας. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε την κατάσταση. Πιο βόρεια έχουμε την Ιουμπάμ Λιβύη, στη Λιβύη. Ένας άλλος τομέας που μας ανησυχεί όλους. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στην περιφερειοποίηση της Αχέλ έχουμε ενσωματώσει και τη Λιβύη, που είναι τμήμα τροποντινά μια περιφερειακή προσπάθεια που δεν περιορίζεται στη Σαχέλ μόνο, αλλά κινείται και πιο βόρεια, λόγω τη παράνομη μετανάστευση και διάφορων συναφών θεμάτων. Για διάφορου λόγου τώρα που ξέρετε καλύτερα από μένα, τους τελευταίους μήνες το πρόβλημα της παράτυπης μετανάστευση έχει μειωθεί κατά τη. Οι που περνούν μέσα από τη Λιβύα. Στην πραγματικότητα έχουμε μετακινηθεί προς τα δυτικά, όμως η προσπάθεια δεν θα μειωθεί για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο εγγύς μέλλον. Η αποστολή κυρίως ήταν στην Τίνιδα, γιατί η Τρίπολη δεν ήταν προσπελάσιμη και δεν μπορούσε να ζήσει κανείς στο παρελθόν. Τώρα όμως έχουμε αυξήσει την παρουσία μας στην Τρίπολη και έχουμε 10 με 12-13 άτομα στην Τρίπολη. Ε, είναι αισθητή η παρουσία μας, είμαστε παρόντες, προσπαθούμε να έρθουμε σε πιο στενή επαφή με τις τοπικές αρχές, με κάποια αποτελέσματα, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μεγαλύτερη ορατότητα για τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέση Ανατολή, άλλε δύο αποστολέ. Η μία είναι πολύ παλιά για την ΚΕΠΑ, η Ιουμπάμα Ράφα. Προς το παρόν ε, δεν μπορεί κανείς να ταξιδέψει τη Ράφα, παρότι πέρυσι πήγαν 10 φορές ε, τα μέλη της αποστολής που ήταν επίτευγμα και η UPOL COPS που συνδέεται περισσότερο με την προετοιμασία και την υποστήριξη της αστυνομίας της Παλαιστινιακής Αρχής ε, με βάση την Ιεριχώ με καλά αποτελέσματα. Ένα από τα καλύτερα της Γιούπολ Cops είναι ότι τη σέβεται και το Ισραήλ. Οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι η αποστολή είναι ένα καλό μέσο διευκόλυνσης των σχέσεων των δυνάμεων του Ισραήλ και των Παλαιστινίων. Με καλά αποτελέσματα λοιπόν. Τελευταία αποστολή. η UAM, η συμβουλευτική αποστολή στο Ιράκ που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο και κάτι. Μικρή αποστολή, αυξάνεται όμως. Έχουμε διπλασιάσει τον αριθμό των μελών της αποστολής. Περίπου 70 άτομα. Θα, φτάσουν, θα, έχουμε 70 άτομα τις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει πρόβλημα λόγω ασφάλειας να έχουμε όλα τα άτομα. Δεν μπορούμε ε, το νέο προσωπικό να το αναπτύξουμε να το έχουμε ας πούμε πριν υπάρχει πραγματικά το πλαίσιο ασφαλεία στο Ιράκ. Και για να έχεις ε, ασφάλεια θέλεις και τεχνικά μέσα και επιμελητιακά μέσα και ανθρώπινους πόρους. Αλλά προχωρούμε. Μας υποδέχονται θετικά οι Ιρακινές αρχές. Υπάρχει πολιτικό πρόβλημα όμως. Ο Υπουργό Εσωτερικών ακόμα δεν έχει διοριστεί ε, και υπάρχει δυσκολία να έρθουμε σε επαφή με άλλες προσωπικότητες ε, του προσωπικού ασφαλείας εκτός Βαγδάτης, όταν αυτή είναι εκτός Βαγδάτης και περιορίζει αυτό το δυναμικό μας. Ε, πιέζουμε όσο μπορούμε σε στενή συνεργασία με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοσφοπέδιο. Είναι η αποστολή που υπέστη τη μεγαλύτερη στρατηγική αναθεώρηση από όλες τις αποστολές. Να σας υπενθυμίσω ότι το 2008 η αποστολή ήταν 3.000 άτομα ε, με εκτελεστικές εξουσίες ε, και στον τομέα του κράτους δικαίου, που ήταν μια νέα προσέγγιση τότε, ήταν η αστυνομία στην πραγματικότητα στο κοσφοπέδιο δύναμη αυτή, ενώ η κοσοβάρικη, αστυνομία ήταν σε εμβριακή φάση και έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Σήμερα Είμαστε στα 500 άτομα, δεν έχουμε εκτελεστικές εξουσίε, ε, ούτε στο επίπεδο του κράτου δικαίου έχουμε εξουσίε. Συνοδεύουμε, συ, Κάποια από τα πιο ευαίσθητα θέματα τα έχουμε παραπέμψει στις ε, τοπικές αρχές πια, τα έχουμε παραδώσει ε, και βοηθήσαμε αυτή τη μετάβαση. Και παρακολουθούμε απλώς από, από τα έξω κάποιες υποθέσεις. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε και το, το ειδικό σώμα ε, που ανήκει στην EULEX, που είναι το ειδικό γραφείο του Ισαγγελέα. έτσι, το οποίο είναι ένα πολύ λεπτό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δικαστήριο αυτό θεωρείται ως δικαστήριο, το δικαστήριο του Κωσφοπεδίου. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αποτελείται από διεθνείς δικαστές και εισαγγελείς και εμείς έχουμε την ευθύνη για το τι θα συμβεί στο εγγύς μέλλον για το δικαστήριο αυτό, το οποίο ξεκίνησε να ερευνά και καλεί ε, κατηγορούμενους για να δώσουν ε, τις ε, καταθέσεις τους ε, στους εισαγγελείς. Έχουν ξεκινήσει, ή ΜΑΝ θα ξεκινήσουν οι ακροάσεις, οι ακροματικές διαδικασίες αργότερα μέσα στο 2019. η αποστολή στην Ουκρανία είναι μια αποστολή που συνοδεύει, είναι αποστολή συμβουλευτική που συνοδεύει την αναδιάρθρωση της αστυνομίας και του κράτους δικαίου. Συμμετείχα στην νομοθετική διαδικασία μαζί με άλλου, γιατί δεν είμαστε εμεί αυτοί που θα ηγηθούμε τη νομοθετική διαδικασία, την υποστηρίζουμε. Έχουμε περιφερειακή παρουσία σε κάποιου τομεί εκτό του Κιέβου, σε κάποιε πόλει. Υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα να επεκταθούμε, αλλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση προ το παρόν και φυσικά η αποστολή ε, επηρεάζεται από τη διαδικασία λήψη αποφάσεων, όπου υπήρχε ο στατιωτικός νόμος που την, ε, που την κήρυξε ο πρόεδρος της Ουκρανίας και η περιστάλη η ελευθερία κινήσεων της αποστολής. Εμείς την περιστήλαμε για να μην δημιουργήσουμε ε, προβλήματα παρεμβολών, ας πούμε, με τους ντόπιου. Τα πάει καλή αποστολή, είναι καλά επανδρομένη, το προσωπικό είναι 100% στο πόσο του, δεν υπάρχουν δυσκολίε καθόλου με τους τοπικούς ομολόγους μας. UM Γεωργία, μετά την UM Ουκρανία. Πάνω από 10 χρόνια είναι εκεί, περιπολούν τα σύνορα, έχουν ε, σημαντικό ρόλο ε, ως διευκολυντές ανάμεσα στους γεωργιανές αρχές και τους Ρώσους και την Νότια Οσετία και διευκολύνουν την ε, διέλευση ε, από την ειδική ζώνη διέλευσης. Ε, το τελευταίο διάστημα σχεδόν όλα τα σημεία διέλευσης έκλεισαν, τα συνοριακά σημεία διέλευσης έκλεισαν, διευκόλυναν όχι μόνο την ανθρωπιστική εκένωση, αλλά και την ιατρική εκένωση, αλλά και δυνατότητα οι φοιτητέ να περάσουν τα σύνορα για να πάνε στα σχολεία. Από τη Δευτέρα άρχισε ξανά το σχολικό, ε, άρχισαν οι να λειτουργούν ε, των ε, έχουμε ένα μηχανισμό και όταν χρειαστεί καλούμε, ερχόμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές, με τις αρμόδιες αρχές για να βρούμε τη λύση. Αυτά τα εργαλεία τα έκλεισαν, παρεμπόδισαν τη λειτουργία του οι για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν συμμετείχαν. Τώρα όμως έχουμε ξανανοίξει αυτή τη δυνατότητα και επομένως λειτουργεί καλά αυτή η αποστολή. Um, Αυτά συνοπτικά ε, σε ό,τι αφορά τις αποστολές επιτόπου και το τι συμβαίνει γύρω από αυτές. Τώρα, τι κάνουμε σε κεντρικό επίπεδο, στις Βρυξέλλες. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν ενεργά παρά το γεγονός ότι θα μπορέσουν να ενισχύσουν τις ε, δεσμεύσεις τους ε, ως προς τις αποστολές και ε, ο λόγος είναι διότι προτιμάμε να έχουμε αποσπασμένους υπαλλήλους εκεί. Προτιμάμε λοιπόν από σπασμένους υπαλλήλου από κάποιο κράτος παρά να γίνονται προσλήψεις επιτόπου. Αυτό εξάλλου βρίσκεται και στην συμφωνία. Επίσης, θα θέλαμε να ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επανεξετάσει τον ε, δημοσιονομικό κανονισμό, τις ε, δημόσιες συμβάσεις, διότι πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόσουμε την νομοθεσία για τις ε, δημόσιες συμβάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι συνθήκες της Βρυξέλλας είναι τελείως διαφορετικές με τις συνθήκες στο πεδίο. δεν είναι το ίδιο το Μπαμάκο, το Μογκαντήσου με τις Βρυξέλλες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε ε, την πραγματικότητα. Δεν θέλω να πω πως ε, πρέπει να μην ακολουθούμε κανέναν κανόνα, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει αρκετή ευελιξία, τουλάχιστον στη διεξαγωγή επιχειρήσεων, διότι χρειάζεται χρόνος μέχρι να αναπτυχθεί, να προετοιμαστεί κάποια επιχείρηση αν ακολουθήσουμε την ε, φυσιολογική οδό, αλλά πολλές ε, φορές χρειάζεται να λάβουμε μέτρα αμέσως. Σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν εσωτερικά, ε, όμως χρειαζόμαστε οπωσδήποτε πόρους οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι και ανα πάσα ε, στιγμή. Ε, σίγουρα είναι δύσκολες οι εποχές και Νομίζω πως ε, ανέλαβα καθήκοντα σε μια εποχή όπου έχουμε όμως και πάρα πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες. Έχω ένα εξαιρετικό επιτελείο στην υπηρεσία μου. Έχουμε τον, ε, την ε, νέα επιτελάρχη η οποία όπως και εγώ παρακολούθησε τις εξελίξεις από την αρχή και νομίζω πως έχουμε αλλάξει αρκετά, αλλά ορισμένες φορές υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται αλλαγή, διότι έχουν λειτουργήσει πάρα πολύ καλά στο παρελθόν. Ε, ίσως μια διαφορετική προσέγγιση. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, διανύουμε περίοδο αλλαγών. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις δράσεις που αναλαμβάνουμε και πρέπει να υπενθυμίζουμε πάντα στον εαυτό μας ότι οι υπηρεσίες που παρέχουμε στο μη στρατητικό σκέλος της CMPD είναι υπηρεσίες που θα δώσουν ασφάλεια και εάν αυξήσουμε τις ε, ικανότητες στην ασφάλεια σε χώρες όπως ε, τη Λιβύη, τη ζώνη του Σαχέλ, στο Κωσυφοπέδιο ακόμα και άλλες, γνώμη μου είναι πως ενισχύεται η συνολική ικανότητα ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώ αντιμετωπίζοντα ε, κάποια προβλήματα που βρίσκονται μακριά από την επικράτειά μα. Οφείλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε την δράση σε αυτούς τους νευραλγικούς τομείς κινητοποιώντας ε, τους αναγκαίους πόρους και φυσικά χρειάζεται σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας έντονη πολιτική στήριξη. Χρειάζεται η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα από τον ε, αριθμό, για παράδειγμα, των, ε, του ανθρώπινου δυναμικού που πρέπει να διαθέσουμε. Αυτά προς το παρόν. Θα σταματήσω εδώ για να μην μακρηγορήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πράγματι ήρθατε στην κατάλληλη στιγμή και επίσης ε, δεν είστε μόνο εσείς τυχαίως αλλά και τα θεσμικά όργανα τυχερά που έχουν εσάς. Θα ε, δώσω τώρα τον λόγο στον ε, Μίχαλ Γκάλερ. Μέχρι τις 3 και 4 έχουμε χρόνο για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή. Και η CPCC όπως και οι άλλοι θεσμοί που έχουμε δημιουργήσει επιφέρουν προστιθέμενη αξία. Είναι μια διτή προσέγγιση με στρατιωτικό και μη στρατιωτικό σκέλος, η οποία καλύπτει περιπτώσεις σε χώρες οι οποίες ε, βρίσκονται σε κρίση, στις οποίες υπάρχουν ένοπλες ε, σειράξεις και φυσικά υπάρχουν προβλήματα είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε όλοι για τα πάντα, αλλά στο μη στρατιωτικό σκέλος πιστεύω πως θα χρειαστεί να παράσχουμε το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και σίγουρα το περιφερειακό επίπεδο είναι ένα επίπεδο στο οποίο χρειάζονται πόροι, το ξέρω και από τη Γερμανία, όπου υπάρχουν αυτά τα τρία ξεχωριστά επίπεδα διακυβέρνησης. Και υπάρχουν πάρα πολλές αποστολές που τρέχουν αυτή τη στιγμή και αν κοιτάξουμε με μεγαλύτερη προσοχή θα δούμε ότι υπάρχουν αρκετές ελλείψεις στην πράξη από αυτά που έχουν συμφωνηθεί στις Βρυξέλλες. Και νομίζω πως ε, οφείλουμε να δώσουμε τη δόση προσοχή εκεί που πραγματικά χρειάζεται και όχι στην θεωρία. Κάτι που σκέφτηκα είναι το εξής. Βλέπουμε ότι έχουμε αυξήσει τον ε, προϋπολογισμό της Frontex. Σίγουρα όχι όσο θα ήθελε η ίδια υπηρεσία, αλλά έχει αυξηθεί ο περιπολογισμό. έχουν γίνει αποσπάσεις από τα κρατη στην ε, Frontex. Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν θα ήταν δυνατόν να δανειστούμε εντό εισαγωγικών προσωπικό από τη Frontex για ε, την CPCC. Ε, αν θα ήταν εφικτό λοιπόν κάτι τέτοιο. Ακριβώς για να αποκτήσουμε το καταρτισμένο προσωπικό που χρειάζεται. Και όχι μόνο από τη Frontex, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ας πούμε, έχει υπαλλήλους οι οποίοι είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Μπορεί να μην χρειαστεί ας πούμε από τα κράτη-μέλη να αποσπάσουν προσωπικό για να βουλώσουν τις τρύπε που έχουν δημιουργηθεί εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα προσθέσω τα εξής και ο Μιχαήλ και εγώ ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στην ε, ε, Γεωργία και επίσης ε, παρακολουθούμε και την δουλειά που γίνεται στην Απχαζία και γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη δέσμευση όσον αφορά τις ε, χώρες αυτές ε, και ε, ότι προχωρούν τα πράγματα. Να σχολιάσω ορισμένα από αυτά που είπατε. Μας είπατε λοιπόν ότι ένα σημαντικό στοιχείο των αποστολών είναι η ποικιλομορφία και βεβαίως αυτό προϋποθέτει και ιδιαίτερες ε, ε, ικανότητες ε, διαχείρισης. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια περισσότερα γι' αυτό και πώς θεωρείτε ότι καλύπτονται ή μπορούν να καλυφθούν οι προκλήσεις που παρουσιάζονται όσον αφορά τη διαχείριση. Επίσης, το θέμα των δημοσίων συμβάσεων ε, υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά την ε, γραφειοκρατία ε, που πρέπει να ξεπεραστεί. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις με τη σειρά που υποβλήθηκαν. Καλύτερη, μεγαλύτερη δέσμευση των κρατών μελών όσον αφορά το compact. Θα είμαι σαφής και χωρίς περικοκλάδες. Υπάρχει δέσμευση, αλλά μερικές φορές πρέπει να έχουμε και αξιοπιστία. Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Λέμε ότι πρέπει να είμαστε σαφείς όταν μιλάμε για το προσωπικό. Να υπενθυμίσω ότι οι αστυνομικοί δεν έχουν ε, ε, ε επιφυλακή, δεν έχουν ε, ε, κάποιες γραμμές ή κάποιους ε, στα μετόπιστε να πούμε ε, είναι όλοι οι καραμπινιέροι π.χ. στην Ιταλία βρίσκονται επί τόπου και στα σημεία δράσης αυτό δεν υπάρχει κανένα αποθεματικό ας πούμε επίσης ε, 27, το συγγνώμη, 28 χώρες μέλη. Βλέπω πολύ, βλέπω πολύ γρήγορα το μέλλον. Ναι, ναι, 28, 28, ζητώ συγγνώμη, είναι λάθος. Εκ παραδρομής έχουμε 28 χώρες μέλη και ενδεχομένως 50 διαφορετικούς τρόπους ε, διαχείρισης ε, των εθνικών εννοείται αστυνομικών δυνάμεων εμείς ε, και από τη δικιά μου χώρα που ξέρω έχουμε αστυνομία, έχουμε καραμπινιέρους, έχουμε σώματα διάφορα. Ε, το ζήτημα είναι χρησιμοποιούν ε, το προσωπικό ή θα χρησιμοποιηθεί το, σωστό, το, το προσωπικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τους σωστούς όρους σύμφωνα με την εντολή. Αυτές είναι ερωτήσεις που εμείς ε, από τις Βρυξέλλες θα πρέπει να απαντήσουμε για να είμαστε αξιόπιστοι και έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να, είναι, να, να δείχνουν πραγματικά εμπιστοσύνη ε, όσον αφορά το προσωπικό το οποίο στέλνουν. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο το οποίο προσπαθούμε τώρα να αποσαφηνίσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Δηλαδή ο τρόπος που επιλέγουμε το προσωπικό να είναι σαφέστερος, ο τρόπος που ε, διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε το προσωπικό επιτόπου να είναι πιο ε, σαφής και αποτελεσματικός. Ε, Γενικώ βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και θα στέλνουν με μεγαλύτερη ευκολία το προσωπικό. Απ' την άλλη πλευρά, ναι, είναι γεγονός ότι πρέπει να δούμε και το διαφορετικό ε, το, το, το διαφορετικό background που μπορεί να έχει ο καθένας ε, στη χώρα του. Τώρα, ε, υποστήριξη από, τις, από τα θεσμικά όργανα, ναι, μπορεί να γίνει και να σας πω ότι Τα συζητούσαμε αυτά και σε μια συνεδρίαση στην ε, δικιά μου, στο δικό μου γραφείο τα συζητούσαμε. Εγώ έχω δέκα αποστολές Έχουμε ανθρώπους που έχουν εξειδίκευση στις δημόσιες συμβάσεις, στα χρηματοπιστωτικά. Η Κομισιόν ξέρει ακριβώς τους κανόνες και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να υποστηριχθούν οι αποστολές από διαφορετικές σκοπιές. Μπορώ να έχω κάποιον από, από μέσα, ε, θα συζητηθεί το θέμα με τους αρμοδίους ε, στην Κομισιόν και βεβαίως ε, θα πρέπει να δούμε τι είδους εμπλοκή θα σήμαινε αυτή, ε, για αυτούς. Αλλά δεν είναι αδύνατον. Συνεργασία χωρίς δομές συγκεκριμένε. Είχαμε, είχαμε ένα αίτημα από την Frontex να βοήθεια για να καθορίσουν καλύτερα ε, την διαδικασία επιλογής προσωπικού και εμείς ε, τους δώσαμε την πραγματογνωμοσύνη μας. Δεν ξέρω πώς θα τη χρησιμοποιήσουν, πάντως έγινε ένα βήμα προς τα εμπρός ε, και υπάρχει λοιπόν μία διάδραση που δεν υπήρχε πριν. Ας δούμε τι μπορεί να γίνει, ας δούμε τι μπορεί να προκύψει στο εγγύς μέλλον και οποτεδήποτε ε, η Frontex χρειάζεται την ε, υποστήριξη ε, για μια αποστολή να δίνεται αυτή η υποστήριξη. Τώρα, όταν μιλάμε για εμπλοκή σε μια αποστολή μακροχρόνια, είναι κάτι διαφορετικό και θα πρέπει να το ξαναδούμε. Τώρα, διαχείριση των αποστολών. Κάθε αποστολή ε, τη διαχειρίζονται οι επαγγελματίες. Αυτοί δηλαδή που έχουν τις επαγγελματικές ικανότητες, που κατανοούν ε, την αποστολή και την χώρα στην οποία ε, θα δουλέψουν. Να σας πω ότι η CPCC δεν παίζει συντονιστικό ρόλο. Εμείς είμαστε το μη στρατιωτικό Operation and Command και συνεχίζω να δίνω ε, κάποιες ε, συμβουλές, ε, οδηγίες, για να μην πω διαταγές, ε, στις αποστολές. Και βεβαίως εγώ έχω και το όλο το υποστηρικτικό μου προσωπικό, το οποίο με ενημερώνει, μου κάνει προτάσεις. Αλλά υπάρχουν αρχές διοικητικές που πρέπει να ακολουθήσουν έτσι ώστε να κάνουν την καλύτερη δυνατή διαχείριση της αποστολής. Ε, ε, η διαχείριση των αποστολών είναι κάτι που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που κάνουμε τώρα. Ναι, φυσικά και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και να σας πω ότι η διαχείριση των αποστολών μέχρι τώρα είναι ε, καλή. Τα οικονομικά. Όσον αφορά τους πόρους, πρέπει να πω ότι οι πόροι που χρειαζόμαστε υπάρχουν είναι εκεί. Και πριν ε, μερικές φορές έχουμε πρόβλημα όταν σε πολύ εξειδικευμένες καταστάσεις πρέπει να εφαρμόσουμε τους γενικούς σηματοδοτικούς κανόνες ε, που ε, μερικές φορές δεν είναι καλά προσαρμοσμένοι στις τοπικές ε, ιδιαιτερότητες. Ειδικά με τις δημόσιες συμβάσεις έχουμε συχνά πρόβλημα. Οι κανόνες μπορεί να είναι εξαιρετικοί και απόλυτα αποδεκτοί για την Ιταλία, για τη Γαλλία, αλλά εδώ θέλουμε να τους εφαρμόσουμε σε χώρες όπου δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής τους. Άρα εκεί χρειάζεται και κάποια ευελιξία και μπορούμε να διαπραγματευτούμε δούμε ε, κάποιο περιθώριο ευελιξίας, το οποίο δεν είναι όμως πολύ μεγάλο. και προσπαθούμε στο κατάλληλο επίπεδο να, ε, και με τις κατάλληλες συνέργειες να προσπαθήσουμε να βρούμε μια διέξοδο. Βεβαίως αυτό δεν είναι πάντα ε, το καλύτερο και δεν γίνεται πάντα. θέλουμε να έχουμε κάτι σαν κανόνα ευελιξίας που μας δίνει όπως σας είπα κάποια ευελιξία σχετική αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να δημιουργηθεί κάποια κρίση ας πούμε. Δεν ξέρω αν απήντησα, βεβαίως απαντήσατε λέει η Πρόεδρος, ε, πάρα πολύ ε, υποβοηθητικά όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Σας ε, διατηρούμε στην ε, πλατφόρμα και προχωράμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Θα ζητήσω από τον ομιλητή του επόμενου σημείου να έρθει. για να συζητήσει ακριβώς αυτό που απασχολεί τον Μίχαελ, ε, τον ρόλο των εθνικών αρχών ε, στις, ε, και των, εθνικών αστυνομικών αρχών κλπ. στις αποστολές ΚΕΠΑ. Perhaps before you start, just on, on, just as you, if I may. Uh, Επιτρέψτε μου. Για τη Λιβύη, για την οποία μιλήσατε. Έχουμε μόνιμη παρουσία, όπως είπατε, με κάποια άτομα εκεί. Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά με δεδομένες συνθήκες που υπάρχουν στη Λιβύη, γιατί ξέρω πόσο γλυπτή είναι η κατάσταση Ε, σε πολιτικό επίπεδο δραστηριοποιούμαστε με την κυβέρνηση, έχουμε τα μέσα για να είμαστε σίγουροι ότι οι άλλοι στην Ανατολή ή όπου είναι τέλο πάντων ε, θεωρούν ότι είναι χρήσιμη αυτή η παρουσία ή απλώς εκτιμούμε τι ρόλο παίζει η σημερινή κυβέρνηση η οποία δεν ελέγχεται καν την πρωτεύουσα. Πολιτικά το στηρίζω. Αν δεν θέλουμε τους Ρώσους ή τους Κινέζους ή ποιον διάολο να κάθεται εκεί στην νότια είσοδο για την Ευρώπη, εμείς πρέπει να κάτσουμε να, παίξουμε αυτό τον ρόλο. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε τη διαφορά εκεί. Μας δέχονται ή τουλάχιστον μας ανέχονται ή είμαστε σημαντικός εταίρος. Πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο, πολύ σύντομα θέλετε κύριε Κόπολα. <laughs> I mean, whatever, if I got it correctly, I mean... Αν σας κατάλαβα, μας ρωτάτε τι μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. As To reinforce our capabilities. Τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας. πώς να το πω, ομά. Έχουμε κάνει πολλά. Έχουμε, δώσει, έχουμε σπαταλήσει πολλούς πόρους. Όταν ξεκίνησαμε την πρώτη αποστολή, και θα το θυμούνται οι προκατοχοί μου. Δεν είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε αυτή την αποστολή γιατί δεν υπήρχε ούτε σχεδιασμό, ούτε έγγραφα, δεν υπήρχε τίποτα, ένα χαρτί γραμμένο, ας πούμε, για να ξεκινήσει η πρώτη αποστολή. Αλλά μέσα σε ένα χρόνο αναπτύχθηκαν δύο αποστολέ. Κάναμε πάρα πολλά έκτοτε. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Η συμμετοχή των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός συνάολων της, ήταν η κινητοποίηση λοιπόν ημών και των κρατών μελών ήταν τεράστια. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Φυσικά μιλήσαμε για κάποια πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε να κάνουμε. Κάποια τουλάχιστον τα έχουμε συμφωνήσει στο χαρτί, ε, μέσω του συμφώνου. Μπορούμε να συνεχίσουμε να τα συζητάμε με τα κράτη-μέλη σε διάφορα επίπεδα, στις Βρυξέλλες και στις πρωτεύουσες πέρσι. Ένας αξιωματικός, ο κ. Πόρτσο, επισκέφθηκε όλες τις πρωτεύουσες και τους υπουργούς ε, εσωτερικών ε, των κρατών μελών για να συζητήσουν τι θα μπορούσε να βελτιωθεί σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των κρατών μελών. Γιατί έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Φυσικά θέλουμε να συνεχίσουμε. Δεν θέλουμε να τα πάρουμε αυτά που κάνουμε πίσω. For, uh, Πάντως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν οι πόροι. Εγώ θα προτιμούσα περισσότερα. Έχουμε το 50% των, του προσωπικού είναι αποσπασμένοι. Φυσικά στις αποστολές υπάρχουν διαφορές. Θα ήθελαμε να έχουμε περισσότερο αποσπασμένο προσωπικό. Για τεχνικούς λόγους ε, θέλουμε αποσπασμένο προσωπικό. Μπορώ να σας πω γιατί. Φυσικά θέλουμε συμμετοχή, έντονη συμμετοχή των κρατών μελών. Αλλά έχουν το απαραίτητο προσωπικό, όπως το ε, Τα οικονομικά δεν είναι πρόβλημα. Ούτε η τεχνική πόρη είναι πρόβλημα. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι λίγο προβληματικό. Δεν έχουμε πάντα τους ανθρώπους που θέλουμε και μερικές φορές υστερούμε και σε ποιότητα. Άρα μπορώ να ζητήσω από τα κράτη-μέλη να στείλουν το καλύτερο προσωπικό που έχουν στη Λιβύη. Ας είμαστε ρεαλιστές. Μπορούν να αποσπάσουν καλά άτομα, αλλά μια χώρα με μεγάλα προβλήματα ασφάλειας θα κρατήσει τους καλύτερους επαγγελματίες στο εσωτερικό της για να λύσει τα δικά της προβλήματα, όχι για να λύσει τα προβλήματα της Λιβύης που είναι μακριά από μας. Αυτές είναι λοιπόν σκέψεις που πρέπει να τις έχουμε υπόψη μας τελικά. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το προσωπικό που έχουμε. Ναι, μπορούμε ή μάλλον θα έπρεπε να πιέσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να μην λησμονούμε ότι πολλή δουλειά έχει γίνει ήδη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θα συνεχίσουμε βέβαια και άλλη φορά ε, το, τη συζήτηση αυτή, ενώ εμείς θα προχωρήσουμε και στο σημείο 9 της ημερησίας διατάξεως, το οποίο αφορά τους ρόλους, το, ρόλο των αστυνομικών δυνάμεων των κρατών μελών στις αποστολές και πά. Μετά έχουμε κοινή ε, ε, συνεδρίαση με μια άλλη επιτροπή στις 4 το απόγευμα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να σταματήσουμε και λίγο πριν από τις 4. Για να προλάβουμε να πάμε στην άλλη αίθουσα. Άρα, άρα Ε, έχουμε ξανασυζητήσει το ρόλο των αστυνομικών δυνάμεων των κρατών μελών και το Compact. Αυτό που θα ήθελα να κάνω τώρα είναι να, να σας παρουσιάσω τον κύριο Κράους Ρέντερ, ο οποίος είναι, προέρχεται από την Δανέζικη αστυνομία, αν δεν κάνω λάθος. Για να μας πείτε πώς βλέπετε τα όσα συμβαίνουν ε, με τις ε, εθνικές αστυνομικές δυνάμεις. Um, and είναι οι τάσεις, ποιες είναι οι συστάσεις ε, που προτείνεται ή θα προτείνεται σε σχέση με τις μη στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και ε, για τα όσα αποτελεσματικά έχετε δώσει όσον αφορά το, το πρόσφατο Compact Agreement. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι μέλη της Υποεπιτροπής, σας ευχαριστώ που δίνετε στην ε, Eurocop, την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Αστομικών Δυνάμεων, για να σας ε, πούνε οι αστομικοί δύναμοι που είναι παρόντες ε, επιτόπου, τις απόψεις τους για τις διεθνείς αποστολές ΚΠΑ και το ρόλο των, ε, των ε, αστυνομικών δυνάμεων. Συγγνώμη. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε αποδεκτά επίπεδα για όλους τους ε, Ευρωπαίους αστυνομικού σε όλες τις αποστολές. Τους δίνει τα εργαλεία και πόρους, ούτως ώστε οι αστυνομικοί να συνεισφέρουν για να προωθήσουν τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και να χτίσουν ε, ισχυρούς τομείς ασφάλειας ε, στις μη στρατιωτικές επιχειρήσεις επιτόπου και να αντιμετωπίσει προκλήσεις της ε, τρομοκρατίας, οργανωμένου κλίματος, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, διαφθοράς. Η αστυνομία είναι βασικό στοιχείο της δημοκρατικής κοινωνίας. Για να πούμε ότι υπάρχει δημοκρατική κοινωνία, πρέπει να υπάρχει αστυνομική δύναμη που να σέβεται το κράτος δικαίου παρά να υπο να υπηρετεί έναν ισχυρό ηγέτη και μπορεί να παρεμβαίνει ε, προς το συμφέρον των πολιτών μόνο υπό, μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο και να, είναι, και να λογοδοτεί. Ε, θέλουμε εμείς ε, να βοηθήσουμε ως Ευρώπη την διεθνή ασφάλεια. Το να υπάρξει μια σταθερή δημόσια τάξη σε αυτές τις χώρες συνδέεται, αυτό συνδέεται με την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σε εμπόλεμες περιοχές όπου υπάρχει στρατιωτική βία και αμέσως μετά τις στρατιωτικές συγκρούσεις. Γι' αυτό ζητάμε ε, να υπάρχουν αποδεκτά πρότυπα που αναγνωρίζουν και την ε, απαιτητική φύση του ρόλου ε, Γι' αυτό γίνεται επαφή των αστυνομικών με τους ψυχολόγους πριν πάνε στην αποστολή και μετά. Οποιοδήποτε αστυνομικό στο εξωτερικό θα πρέπει να πηγαίνει σε τις αποστολές μόνο εφόσον το επιθυμεί. Η ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων στο εξωτερικό δεν συγκρίνεται με την κλασική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στη χώρα του, του χώρα μας. Θα πρέπει οι αστυνομικοί να είναι καλά προετοιμασμένοι για να πάνε στο εξωτερικό για να ξέρουν το περιεχόμενο, να έχουν το ε, εξοπλισμό και να έχουν γνώση της τεχνολογίας και να τους υποστηρίζουμε σε συνεχή βάση. Έχουμε δει στη Eurocop ότι κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να δώσουν κατάρτιση ούτε εκπαίδευση σε αστυνομικούς ε, ε, οι οποίοι βρίσκονται σε, ξένες, σε αποστολές του εξωτερικό. Γι' αυτό θέλουμε ειδική εκπαίδευση για αυτούς τους αστυνομικούς, ούτως ώστε κανένας αστυνομικός να πηγαίνει στο εξωτερικό σε τέτοιες αποστολές χωρίς επαρκή κατάρτιση και χωρίς να ξέρει τα αστυνομικά του δικαιώματα, τα επίσημα δικαιώματά του και τα καθήκοντά του. Αυτό συνδέεται με το ερώτημά σα, αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη Frontex και το προσωπικό τη Frontex σε αποστολέ. ΚΠΑ. Κατά την προσωπική μου άποψη και στην CPCC. Θα ήταν πρόβλημα αυτό, γιατί οι αστυνομικοί της Frontex δεν έχουν ε, αυτή την εκπαίδευση πριν ε, από την αποστολή. Δεν έχουν αυτά τα μαθήματα, ας πούμε, προετοιμασίας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Οι αστυνομικοί επίσης θα πρέπει να έχουν και γλωσσική κατάρτιση, ασφαλή συστήματα επικοινωνίας, πέρα από τα πολιτιστικά στοιχεία που αφορούν την περιοχή στην οποία θα πάνε. Φυσικά, το να υπάρχει υψηλής ποιότητας εξατομικευμένος εξοπλισμός, ασφαλές τόπος ξεκούρασης, ε, απολαβές, τόπος διαμονής κτλ. που θα αναγνωρίζει τους κινδύνους της εργασίας στο εξωτερικό και ε, πρόνοια σε περίπτωση ατυχήματος καθώς και στα αξιωτικά δικαιώματα είναι βασικά θέματα αυτά. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μέγιστη ασφάλεια και ε, διασφάλεια, ε, ασφάλεια ζωής ε, που συνδέεται με την αποστολή στο εξωτερικό. Κάθε αστυνομικός θα πρέπει να έχει την ασφάλεια που τον καλύπτει όσον τον περισσότερο. Στη Δανία 2010-2011 ασχοληθήκαμε με ειδικούς Δανέζους αστυνομικούς ε, που πήγαν στο εξωτερικό σε βελτιωμένες συνθήκες. Γιατί κάναμε αυτή την προσπάθεια στη Δανία. Γιατί είδαμε ότι όλο και περισσότεροι αστυνομικοί είχαν ε, επαγγελματικές, ψυχολογικές, ε, ψυχολογικά προβλήματα μετά τις αποστολές που, στις οποίες υπηρέτησαν στις δεκαετίες, στην δεκαετία του 90. Κυρίως είχαν το λεγόμενο μετατραυματικό ε, σύνδρομο. Ε, και χάρη σε, αυτά, σε αυτές τις προσπάθειες φτάσαμε σε καλά αποτελέσματα. Επίσης, δίνουμε ψυχολογική βοήθεια πριν και μετά την αποστολή. Συμφωνήσαμε με τον Αρμόδιο Επίτροπο για τις διεθνείς αποστολές ότι θα πρέπει να μιλήσει ο αστυνομικό ατομικά ε, και εξατομικευμένα πριν, με ψυχολόγο πριν και μετά την αποστολή. Το κάναμε και κάποιες, ε, κάποια τεστ, κάποιες δοκιμές το που ξεκίνησαν το 2013 ε, πριν πάει ο αστυνομικό ε, στην αποστολή. Και όταν τα κάναμε αυτά τα τεστ είδαμε ότι πάνω από το 50% των αστυνομικών δεν πέρασαν αυτά τα τεστ γιατί δεν είχαν αντιμετωπιστεί κάποια ψυχολογικά προβλήματα, υπήρχαν προβλήματα ας πούμε αλκοολισμού και άλλα προσωπικά προβλήματα ε, σε συνάφεια πάντα με τις αποστολές τους και την εργασία τους. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε στην υποχρεότητα των ευρωπαϊκών προτύπων ε, για σε φυσικό και ψυχολογικό επίπεδο για τους αστυνομικούς. Στην Δανία ε, διαπραγματευτήκαμε το Διεθνή ε, Επίτροπο και έχουμε ένα σύστημα μέτρησης ε, που αναπτύξαμε μαζί με ψυχολόγους και εκπροσώπους της Διεθνούς Επιτροπής και εκπροσώπους της Ένωσης για να επισκέπτονται τους συναδέλφους μας μία με δύο φορές το χρόνο ανάλογα με την κατάσταση αποστολής, δηλαδή αν είναι εμπόλεμη ζώνη στο Ιράκ, Φερρυπίν, ή στην, στην ανατολική περιοχή της Ουκρανίας ή σε μια εμπόλεμη περιοχή, Γεωργία, Κοσφοπέδιο. Για να υποστηρίξουν τους αστυνομικούς, να τους βοηθήσουν ε, σε μία συνεχή βάση. Επίσης, υπάρχει μία ομάδα προετοιμασίας ε, για επίγοντα που μπορεί να αντιδράσει πάρα αυτά μέσα σε ώρες, μέρες από την ε, περίπτωση που γίνουν ατυχήματα σοβαρά ή απόπειρα αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια τη αποστολή. Ε, με ψυχολόγο, <coughs> εκπρόσωπο τη Διεθνού Επιτροπή και εκπρόσωπο από την Ένωση. Ε, ε, έχουμε κάνει εμβόλια, διπλωματικά διαβατήρια για τους αστυνομικούς μας, που σημαίνει ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε πολύ γρήγορα μετά την εκδήλωση του προβλήματος και πάρα πολύ συχνά έχουμε χρησιμοποιήσει αυτές τις δυνατότητε, ειδικά όταν είχαμε την ε, ε, αποστολή ΟΙΠΟΛ στο Αφγανιστάν. Επίσης κάναμε και άλλες συμφωνίες. 21 εθνικές συμφωνίες που βελτίωσαν την, ε, τη συνθήκη για ε, των αστυνομικών που συμμετέχουν σε διεθνείς αποστολές. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό η Eurocop να δίνει την άποψή της για τις εργασιακές σχέσεις σε αποστολές για θέματα εργασιακών σχέσεων στις αποστολές ΕΚΠΑ. Η Eurocop ζητά ε, δεσμευτικά πρότυπα για τη συμμετοχή ε, των εκπροσώπων των συνδικάτων των αστυνομικών στα εν λόγω κράτη. για αυτά τα συνδικάτα πρέπει να ε, δημιουργηθούν πάρα αυτά, ούτω ώστε να συναπευθυνθούν, να δούμε ποια είναι τα αρμόδια συνδικάτα σε περίπτωση απόσπασης αστυνομικών. Πιστεύουμε ότι αυτά τα στοιχεία θα εμπνεύσουν και θα εφαρμοστούν στις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑ στα πλαίσια του Συμφώνου και στα εθνικά σχέδια ε, που αναπτύσσουν τα κράτη τα επόμενα χρόνια. Ε, στα εθνικά σχέδια που θα αναπτύξουν τα κράτη τα επόμενα χρόνια. Και να εφαρμοστεί λοιπόν, να εφαρμοστούν όλα αυτά στα πλαίσια του Συμφώνου, του Compact. Τέλος, από τις 10 αποστολές που αναφέρθηκαν έχουμε δανούς αστυνομικού στις μισές και επίσης υπάρχουν και εκπαιδευτές οι οποίοι βοηθούν τις ε, αποστολές αυτές ιδιαίτερα στο Ιράκ. Σας ευχαριστώ πολύ και φυσικά θα δεχτώ τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ρέτεν. Ως ε, πρώην συνδικαλίστρια μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας με την ανάγκη να υπάρχει εκπρόσωπος των ε, συνδικάτων ιδιαίτερα σε τέτοιες ε, περιπτώσεις που είπατε εσείς ε, για να λυθούν διάφορα ψυχολογικά θέματα και να αποτραπούν οι ψυχολογικοί κίνδυνοι και σωματικοί. Όμως, θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο για, στον αντιστράτηγο για κάποια επιπλέον σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Ε, εξηγήσατε πολύ καλά ε, αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά θα προσθέσω σε ό,τι αφορά την κατάρτιση ότι είναι κοινή ευθύνη των ε, κρατών μελών, τα οποία πρέπει να παρέχουν όχι μόνο τους υποψήφιους, αλλά και να τους καταρτίζουν για τις αποστολές στις οποίες θα σταλούν. Φυσικά η διαδικασία επιλογής θα πρέπει να είναι και μετά υπάρχει και η ευθύνη για τις αποστολές επιτόπου. Δεν μιλάμε βέβαια για κατάρτιση δύο, τριών, τεσσάρων ημερών. Η κατάρτιση του προσωπικού πρέπει να είναι συνεχιζόμενη και διαρκής, έτσι ώστε όσοι συμμετέχουν στις αποστολές αυτές ε, να γνωρίζουν τις ε, εντολές, ε, τη διάρκεια της εντολής, τις ευθύνες τους, το τι πρέπει να κάνουν και τη διάρκεια μιας αποστολής. Όλοι λοιπόν έχουν αυτήν την υποχρέωση. Μετά, υποβολή έκθεση σχετικά με την αποστολή. Κάποιες χώρες έχουν μία πιο ενδελεχή διαδικασία, κάποιες άλλες χώρες λιγότερο. Φυσικά υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη, υπάρχει και διαφορετικό σύστημα από χώρα σε χώρα. Ορισμένες χώρες επίσης μπορεί να μην ε, δίνονται ή να μην θέλουν να αλλάξουν το σύστημα, οπότε θα μπορούσαμε να προτείνουμε μεν βελτιώσεις, αλλά δεν μπορούμε να τις επιβάλλουμε. Μετά σε ό,τι αφορά την ε, παροχή βοήθειας, ιατρικής ή ψυχολογικής, στο προσωπικό πριν μια αποστολή. Θα πρέπει φυσικά να γίνεται μια πρώτερη αξιολόγηση, η οποία θα βοηθήσει ε, και στις αποστολές και κατά τη διάρκεια μιας αποστολής πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα παροχής ιατρικής ε, βοήθειας, όχι ψυχολογικής. Όμως, υπάρχουν λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να κοιτάξουμε πώς ακριβώς θα γίνεται η παροχή της ε, ιατρικής βοήθειας, ποιες θα είναι οι λεπτομέρειες. Να δούμε με ποιο τρόπο θα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε τις συστάσεις. Ε, βέβαια αυτό δεν είναι κάτι που θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες ε, σχετικά με τα συνδικάτα, αλλά θα σας πω πως ε, δεν χρησιμοποιούμε μόνο αστυνομικούς αλλά και υπαλλήλου από άλλες υπηρεσίες. Πριν από μία αποστολή. Εδώ βέβαια ισχύουν Ισχύει μάλλον η εθνική νομοθεσία. Υπάρχουν κανόνες που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η αρμόδια αρχή είναι εκείνη που καθορίζει τις λεπτομέρειες μιας αποστολής. Και αυτό φυσικά αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Δεν είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να παρέμβουμε. Φυσικά και μπορούμε να το συζητήσουμε με τα κρατημέλη, αλλά ως εκεί. Και φυσικά θα έπρεπε να υπάρχει ένας εκπρόσωπος ε, της αστυνομίας, ο οποίος έχει λόγο αλλά στην Ιταλία, για παράδειγμα, τα συνδικάτα της αστυνομίας αφορούν την αστυνομία μόνο. Οι καραμπινιέροι ε, προσωπούνται από άλλο φορέα. Υπάρχει εσωτερική διαδικασία σε άλλο επίπεδο εκπροσώπησης. Βέβαια, τα συνδικάτα, ξέρετε, έχουν την τάση να επεκτείνουν τις ε, αρμοδιότητές τους και τις εξουσίες τους και να επεκτείνονται γενικότερα. Οπότε χρειάζεται προσοχή και να αναγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Ωστόσο, να πω ότι υπάρχει μεικτή αρμοδιότητα. Υπάρχει και η εθνική αρμοδιότητα, υπάρχει η κοινή αρμοδιότητα, η ευρωπαϊκή ε, τα λοιπά, Υπάρχουν τα διάφορα θεσμικά όργανα που ε, εμπλέκονται, υπάρχουν τα Ηνωμένα Έθνη. Βέβαια, υπάρχουν και αρκετές γκρίζες ε, ζώνες, ε, τις οποίες δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε. Είναι όμως σημαντικό να εντοπίσουμε ακριβώς αυτές ε, τις ε, περιπτώσεις, διότι υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν έγγραφα τα οποία αναφέρουν με λεπτομέρειες ε, ποιο είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση πριν από μια αποστολή, κατά την αποστολή, τι γίνεται κτλ. Και όλα αυτά, όλοι αυτοί οι κανονισμοί, αυτά τα έγγραφα προϋπήρχαν Είχαμε στείλει στα κρατημέλη της, ε, την ενημέρωση λοιπόν σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν, με το τι κατάρτιση πρέπει να έχει το προσωπικό που θα στείλουν στις αποστολές κτλ. Είχαν όλες λοιπόν τις λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις αποστολές και στην αρχή η συμμετοχή ήταν μόνο των, της αστυνομίας ή κατά 95% αστυνομία. Τώρα φυσικά έχει αλλάξει αυτό, υπάρχουν διάφοροι ε, εργαζόμενοι από πολλούς τομείς που συμμετέχουν σε μια αστυνομική αποστολή και υποβοηθούν το έργο της αστυνομίας. Η UBAM, ας πούμε, στη Λιβύη είναι μια τέτοια περίπτωση. Υπάρχει η EU CAP, η ικανότητες, υπάρχουν οι αποστολές παρακολούθησης, αποστολές ελέγχου. Ε, η κάθε μία αποστολή έχει διαφορετικά καθήκοντα. Μιλώ για τις αποστολές μη στρατιωτικού χαρακτήρα. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Μίχαηλ το άλλο μέλος της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ για τις επεξηγήσεις. Ήμουνα στο CPCC ε, ε, και εσείς αναφερόσαστε στο ε, CSTP. Έχουμε στρατιωτικές και μη στρατιωτικές αποστολές και πάνω. Ε, συμμερίζομαι τα περισσότερα από αυτά που είπατε και σε μεγάλο βαθμό μάλιστα. Και αυτά που προσέθεσε ο κύριος Κόπολα πραγματικά ε, αποσαφηνίζουν και τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπατε ότι υπάρχουν κάποιες χώρες μέλη που δεν είναι σε θέση να ε, ε, έχουν την να παράσχουν την απαραίτητη προετοιμασία. Ρωτώ λοιπόν από πλευρά της Ένωσης, μήπω πριν φτάσουν ε, να αξιολογούμε τι χρειάζονται την ώρα της άφηξής τους, γιατί φαντάζομαι ότι όταν θα γίνει η ανάπτυξη επιτόπου θα είναι λίγο αργά. Υπάρχουν παρατηρητές, παρατηρητές που είναι στη θέση αυτή πολλά χρόνια και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Θα μπορούσα επίσης να φανταστώ ότι εάν η προετοιμασία για την χώρα προς την οποία ε, θα πάτε, ας πούμε στην περίπτωση του Κωσυφοπεδίου, ε, ένας Έλληνας αστυνομικός που θα πάει στο Κωσυφοπαίδιο ίσως θα πάρει διαφορετικές πληροφορίες για το τι συμβαίνει εκεί ε, σε σχέση με κάποιον εστονό συνάδελφό του που θα πάει στο Κωσυφοπαίδιο. Θα πρέπει να δούμε περί τίνος πρόκειται και ε, οπωσδήποτε χρειαζόμαστε και κάποιες ε, ε, mainstreaming συμβουλές ας πούμε ή προετοιμασία. Το ίδιο ισχύει και για το υλικό. Ερώτηση λοιπόν θα πρέπει όλοι να έχουν τον ίδιο εξοπλισμό. Και μάλλον να ρωτήσω, σε αυτές τις αποστολές δίνουμε, παρέχουμε το απαραίτητο υλικό, το απαραίτητο εξοπλισμό, έχουν οι αστυνομικοί πούμε, την υποχρέωση να, φέρουν τα δικά τους όπλα και ε, ξέρουμε αν έχουν όλοι το, τον ίδιο εξοπλισμό. Υπάρχει κάποιο απόθεμα, κάποιο στόκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτού του είδους τον εξοπλισμό όλοι λοιπόν να έχουν ε, τα ίδια εργαλεία με τα οποία θα δουλέψουν επί τόπου. Και επίσης όσον αφορά τους όρους αναφοράς, αυτό που είπατε για τις ε, ε, για την ασφάλεια και για τις ε, συντάξεις και τα συντάξιμα χρόνια κτλ. Ναι, είναι σωστό. Θα πρέπει να υπάρξουν εγγυήσει και τι θα, ε, τι, ποια θα είναι η αποζημίωσή τους εάν έχουν κάποιο πρόβλημα, εάν τραυματιστούν κτλ εγώ είμαι απολύτως υπέρ του να πούμε χρειαζόμαστε κάτι εναρμονισμένο και βεβαίως στο μέγιστο δυνατό ε, επίπεδο γιατί διαφορετικά ε, αν θέλουμε και τα καλύτερα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να μην δώσουμε κι εμείς κάτι. Όταν βρούμε και όταν βρίσκουμε λοιπόν αυτά τα καλά στοιχεία θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να προχωράμε και στην σωστή τους αντιμετώπιση. Kind of Uh, where do we stand? Are Και ρωτώ λοιπόν, είμαστε σε θέση να παράσχουμε ε, τα καλύτερα δυνατά, τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις κτλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μιχαήλ. Ε, τώρα θα υπογραμμίσω πάλι ότι δεν ε, έχουμε χρόνο. Ξέρω ότι είναι άδικο αυτό, αλλά θα πω και εγώ δύο λόγια όμως έχουμε ε, την ε, ΣΥΠΧΟ, ε, την, αστυνομική, την Ενωσιακή Υπηρεσία για την Κατάρτιση των Αστυνομικών. Εκεί θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία. Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω και το θέμα το οποίο ανέφερε ο μιλτής προηγουμένως όταν κάνει λόγο για την ιατρική υποστήριξη του προσωπικού που βρίσκεται σε αποστολή και ε, εγώ δεν θα ήθελα να πούμε ε, την ιατρική υποστήριξη και ψυχολογική υποστήριξη. Θα ήθελα η ψυχολογική υποστήριξη να ε, βρίσκεται εντός, να συμπεριλαμβάνεται στην ιατρική περίθαλψη. Έχετε πέντε λεπτά το πολύ. Σας το λέω. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με αυτό που είπατε εσείς, δηλαδή ότι η ψυχολογική υποστήριξη θα έπρεπε ε, να είναι ε, μέρος της ε, ιατρικής υποστήριξης. αλλά ξέρετε, καμιά φορά. Πολύ συχνά ο αστυνομικό που αντιμετωπίζει προβλήματα θέλει να μιλήσει με κάποιον που μιλάει τη δικιά του γλώσσα για, τους, για τις στολές. Εγώ δεν αναφέρομαι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, λέγοντας ότι δεν, ε, δεν προσέχουν ας πούμε τους αστυνομικούς και τον εξοπλισμό τους. Εγώ λέω απλώς ότι όταν πηγαίνουν σε εξωτερικές αποστολές θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τον εξοπλισμό. Δεν είναι το ίδιο να πας στο Μαλί ε, και στην Ανατολική Ουκρανία όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατεβεί στους μείων 15 ε, βαθμούς Κελσίου. Λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα standard package και μετά, και μετά τα εξειδικευμένα στοιχεία για την κάθε αποστολή. Σε μερικέ χώρες τα πράγματα είναι καλά, σε άλλες χώρες όμως μπορούν να βελτιωθούν πολύ εμπνεόμενοι από τις χώρες όπου τα πράγματα πάνε καλά όσον αφορά την πίεση στις εθνικές αστυνομικές δυνάμεις. Θα συμφωνήσω απολύτως με τον κύριο Κόπολα. Πρέπει να δούμε πώς είναι η κατάσταση επιτόπου σε σχέση ας πούμε με την ε, ε, μεταναστευτική κρίση, το προσφυγικό. Μερικές φορές όντως λείπουν και οι κατάλληλα ε, προσοντούχοι ετούντες. Γι' αυτό μεταξύ των προτάσεων που έκανα, εάν θέλει κανείς να γίνει μέλος του top management, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να πας σε διεθνείς αποστολές, ε, έτσι ώστε να το βάλεις στο βιογραφικό σου κατά κάποιο τρόπο, να ξέρεις και μετά έχει ε, βεβαίω ε, μεγαλύτερε πιθανότητε για γίνεις top manager στην αστυνομία. Όσον αφορά τι ασφάλειες. δεν ε, συμβαίνει αυτό σε όλες τις χώρες. Σε μερικές χώρες δηλαδή υπάρχουν προβλεπόμενες ασφάλειες. Το θέμα είναι αν θα καταφέρουμε να ε, πείσουμε τις χώρες οι οποίες υπολείπονται ε, να αυξήσουν το επίπεδο. Σύμφωνα απόλυτα με τον Κλάους. να προσθέσω κι εγώ κάποια πράγματα. Οι ασφάλειες λοιπόν υπάρχει ασφάλιση για τους ε, αστυνομικού που συμμετέχουν σε μια αποστολή και πρέπει να υπάρχει βέβαια και τρόπο οικονομική κάλυψης αυτή τη ε, ασφάλιση. Σίγουρα είναι ασφαλισμένη η αποστολή, όμως είναι καλό και ο αστυνομικό να ξέρει ότι είναι ασφαλισμένο από το εθνικό του σύστημα ε, σε περίπτωση που ομιγέννητο συμβεί κάτι άσχημο, χάσει τη ζωή του ως αστυνομικό, ότι θα είναι εξασφαλισμένη η οικογένειά του. Και πάλι κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες και το θέμα ε, είναι αν μπορούμε να πιέσουμε τα κράτη-μέλη για να αναθεωρήσουν τις πρακτικές τους. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε κάποια σύσταση, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Συνήθως τώρα, σε ό,τι αφορά την εξάρτηση, τους ε, παρέχουμε Φραγιλέκα, ε, ασύρματους, ε, μέσω επικοινωνίας, τους παρέχουμε διάφορα και φυσικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους στολές και μπορούν να έρθουν με το δικό τους όπλο. Και γιατί είναι σημαντικό να έχουν τα δικά τους όπλα, διότι πάνω σε αυτά εκπαιδεύτηκαν. Επίσης υπάρχουν και ομάδες security οι οποίες παρέχουν ασφάλεια σε όσους δεν είναι σε θέση να ε, στήσουν ας πούμε τους ε, φράχτες. Όλα αυτά τα παρέχει αποστολή. Και οι φρουροί, οι σωματοφύλακες ας πούμε και όλοι έχουν, χρησιμοποιούν υλικά που παρέχονται από την αποστολή αλλά και ε, καταρτίζονται από προγράμματα της αποστολής. Και φυσικά υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα όσα δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα όσα δίνουν τα κρατημέλη. Κάποιοι δίνουν περισσότερα, κάποιοι λιγότερα. Ωστόσο, δίνεται μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια, στην ιατρική φροντίδα και όπως είπε πολύ σωστά ο Κλάους πρέπει κανονικά η ψυχιατρική βοήθεια, η ψυχολογική βοήθεια να θεωρείται ιατρική βοήθεια και φυσικά αν χρειάζομαι ψυχολογική υποστήριξη θα πρέπει να έχω το δικαίωμα να το κάνω στη γλώσσα μου. Διότι αν μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα σίγουρα μπορώ να μιλήσω με περισσότερη ακρίβεια από ότι αν μιλήσω γαλλικά ή αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ε, μη στρατιωτικέ αποστολές. Και σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας και στο πρώτο πάνελ. Εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτού του μέρους της συνεδρίασης της Επιτροπής ΣΕΝΤΕ. Τώρα θα πάμε στην αίθουσα 3G3, δηλαδή δύο ρόφους πάνω. Σε τρία λεπτά ξεκινάμε. Thank you.